Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Ε, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Τομπίας Φλούγκερ γνωστοποίησε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον της εισαγγελίας Μονάχου. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 του κανονισμού, η αίτηση αυτή διαβιβάστηκε στην αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Τώρα ερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη, η οποία προβλέπει τις προφορικές ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τους ίνους ροζέ και τις επιτρεπόμενες ινολογικές πρακτικές. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες που θα πάρουν το λόγο. Πρώτη έχει το λόγο η κυρία Λούλινγκ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η παραγωγή ίνων ποιότητος, αλλά και οι ευφυείς καταναλωτές, αυτοί οι οποίοι είναι γευσιγνώστες και γνωρίζουν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, δεν θέλουν να ακούνε για ίνους από ανάμειγμα.